My αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσω με τους παρόντες. Αλλιώς θα ξεμείνουμε από χρόνο και θα πρέπει στις 10.45 ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, έχουμε την κοινή συζήτηση και την όλη παρουσίαση για, για την πολιτική όσον αφορά τα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κυρία Σπινάντ της Γενικής Διευθύνσεως Δικαιοσύνης θα μιλήσει για το θέμα των ναρκωτικών. Ε, θα κάνει μια εισαγωγή στο θέμα και ποια είναι όλη η κατάσταση της πολιτικής κατά των ναρκωτικών και τις διάφορες εξελίξεις. Και έχουμε την παρουσία του κυρίου Γκέτς, του Διευθυντού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας ο οποίο θα παρουσιάσει τη γενική έκθεση του Φορέα για το 2012 και το πρόγραμμα εργασιών για το 2013-2015. Λοιπόν, καταρχάς θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στον κύριο Γκέτς και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Σαλβατόρε, αγαπητέ Βόλφκανγκ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλη των θεσμικών οργάνων. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που συμμετέχω σήμερα σε αυτή τη συζήτηση για το πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της πλέον πρόσφατης εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Ε, αυτή η έκθεση από τον φορέα αυτό είναι μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών και ανάλυσης ε, είναι πολύ ψηλή και πλήρη ανάλυση όσον αφορά την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μα βοηθά όλου να κάνουμε παίρνουμε εμπεριστατωμένε αποφάσει και να δημορφώνουμε τι κατάλληλε πολιτικέ για τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βόλφκανγκ θα δώσει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία και τι τάσει όσον αφορά τα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πω στα γρήγορα δύο λόγια για το θέμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντα ότι παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφύγει κάποια από τα χειρότερα προβλήματα που κάποιες χώρες και περιοχές του κόσμου αντιμετωπίζουν λόγω των παράνομων ναρκωτικών, όπως επιδημίες AIDS, λόγω χρήσεως ενέσεων για ναρκωτικά ή ε, προβλήματα χωρών που παράγουν ναρκωτικά ή που κυκλοφορούν τα ναρκωτικά. Η προβληματα χωρων που παραγουν έχει σταθεροποιηθεί μεν τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξακολουθεί να είναι πρόβλημα περίπλοκο υγεία και κοινωνικό πρόβλημα που πλήττει εκατομμύρια Ευρωπαίου. Σκεφτείτε και μόνο ότι σε αυτή τη μία ώρα τη εξαγωγή τη συζητήσεω ένα άνθρωπο θα πεθάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω υπερβολική δόση ναρκωτικών. Πιθανότατα θα είναι και κάποιο νέο. Ε, σκοτώνεται ε, ένα άτομο κάθε 8.000 άτομα το χρόνο που πεθαίνουν. Και σήμερα, μόνο σήμερα, η παράνομη, το παράνομο εμπόριο θα αποδώσει 200 εκατομμύρια περίπου ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα παράνομα δίκτυα κυκλοφορίας ναρκωτικών. Διότι αυτό είναι το προϊόν. Ο πλούτος που παράγεται από τα ναρκωτικά είναι περίπου 70 δις ευρώ το χρόνο. Αυτά τα χρήματα δίνουν τη δύναμη στα δίκτυα κυκλοφορία εμπορίου των ναρκωτικών, μπορούν να επενδύουν ε, σε πάρα πολλού τομεί, δραστηριότητε παράνομες και νόμιμε, και όλα αυτά υπονομεύουν την ασφάλεια των ε, οικονομιών μας. Κυρίε και κύριοι, ε, γνωρίζουμε ότι η μετώπιση του προβλήματος απαιτεί μακροπρόθεσμη, ολοκληρωμένη και πολυτομιακή προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναρκωτικά παρούσες στατικικές εκπνέουν στο τέλος του έτους και με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι την περασμένη εβδομάδα επετεύχθη μια συμφωνία σε επίπεδο ομάδων εργασία για νέα στρατηγική ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2020. Αυτή η στρατηγική των ναρκωτικών βασίζεται στα επιτευχθέντα στις πολιτικές ναρκωτικών στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Ε, φτάσαμε σε μια συμφωνία χάρη στις μεγάλες προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας και αναμένεται το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνουν την αισθητική τα ναρκωτικά τις επόμενες εβδομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστηρίξει πλήρω την Κυπριακή Προεδρία για την επίτευξη συμφωνία επί μια στρατηγική. Καταρχά ξεκίνησε και υποστήριξε ανεξάρτητη αξιολόγηση ε, της, ε, των, των στρατηγικών που εφαρμόζουμε τώρα. Και από αυτών των στρατηγικών βασίζεται η νέα στρατηγική. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Σαλβατόρε Γιακολίνο, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην αξιολόγηση στατικής των ναρκωτικών ως μέλος της ε, διευθύνουσας ομάδας όσον αφορά την αξιολόγηση στρατηγική εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η συμμετοχή του στι συζητήσει ε, μα ενέπνευσε τα μάλα. Ε, η νέα στρατηγική των ναρκωτικά οικοδομείται στο ευρωπαϊκό μοντέλο για τα ναρκωτικά, όπω είναι γνωστό. ακολουθούμε ισορροπημένη πολιτική για τα ναρκωτικά, άρα πρέπει εξίσου να αντιμετωπίζουμε και τη ζήτηση και την ε, ε, προμήθεια ε, ναρκωτικών. Δηλαδή η ζήτηση και η προσφορά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού διότι επηρεάζουν τον ατάλλο. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε πολιτικές που βασίζονται επί συγκεκριμένων, δηλαδή θέλουμε επιστημονικά στοιχεία και επ' αυτόν βασίζουμε τις πολιτικές που επιλέγουμε και εδώ ο ρόλος του παρατηρητηρίου είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μας δίνει τα κατάλληλα στοιχεία για να μπορούμε να κάνουμε περιστατωμένες ε, κινήσεις. Αυτή η στατική ναρκωτικά θα παίξει θεμελιώδη ρόλο ούτω ώστε να ακολουθούμε συνεκτική προσέγγιση σε όλου του τομείς πολιτική που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για αποτελεσματική πολιτική για την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Χρειάζεται σύγκληση μεταξύ των πολιτικών των κρατών μελών για τα ναρκωτικά και χρειάζεται και συνέπεια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δράσεων για τα ναρκωτικά. Η στρατηγική θα εφαρμοστεί μέσω δύο διαδοχικών σχεδίων δράση για τα ναρκωτικά που θα καθορίζουν πολύ συγκεκριμένε δράσει που θα πρέπει να αναλυθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με την Ιρλανδική Προεδρία που θα ακολουθήσει Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα συντάξει το πρώτο σχέδιο δράσης, εφαρμοστικό σχέδιο δράσης. Να σας πω εν ολίγης ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ναρκωτικά και ποιο είναι το πρόγραμμα για τα ναρκωτικά που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ναρκωτικά θα παρουσιαστούν σε μια ανακοίνωση για ισχυρότερη απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ναρκωτικά που θετήθηκε προ έτου έτους ακριβώς τον Οκτώβριο του 2011. Αυτή η ανακοίνωση ε, δημιουργεί τη βάση και το σκηνικό για την πλήρη αναθεώρηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά και του σχετικού πλαισίου. Πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκε η ενίσχυση των νομοθετικών προτάσεων όσον αφορά νέες ψυχοδραστικές ε, ουσίες ψυχοτρόπες ουσίες και το νομοθετικό πλαίσιο για το εμπόριο των ναρκωτικών, τα σχετικά δικήματα και τις ποινικέ κυρώσεις. Την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την χρήση των πρόδρομων ουσιών για τα ναρκωτικά. Και ανακοίνωσε επίσης την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την κατάσχεση ανάκτηση πόρων και καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, παρανόμων εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα χρόνο αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει παρουσιάσει τις μισές από αυτές τις νομοθετικές προτάσεις. Τον Μάρτιο υπέβαλε νομοθετικές προτάσεις για κατάσχεση και ανάκτηση πόρων και οι συνάδελφοι από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση θα σας μιλήσει περισσότερο αργότερα για το θέμα αυτό. Τον Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε δύο νομοθετικές προτάσεις για την ενίσχυση των κανόνων που μας βοηθά να καταπολεμήσουμε την χρήση των προδρόμων ουσιών, χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων, νομικών ουσιών, μπορεί να χρησιμοποιηθούν νόμιμα, αλλά χρησιμοποιηθούν κακώς για την παράνομη παραγωγή ναρκωτικών ουσιών. Και οι τρεις άλλες νομοθετικές προτάσεις ανακοινώθηκαν και αυτές στην ανακοίνωση και έχουν δρομολογηθεί, είναι καθοδόν και θα παρουσιαστούν πιθανότατα τους ε, επόμενους μήνες. Καταρχάς, η πρώτη νομοθετική πρόταση αφορά τις νέες ε, ψυχότροπες αυτές, ψυχοτροπικές ουσίες. Αυτές είναι για προτεραιότητα για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για σας, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα τα πολλά κοινοβουλευτικά ερωτήματα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις νέες ουσίες και οι ερωτήσεις μας αφορούν το τι σκοπεύουμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο για το ζήτημα αυτό και θέλουμε ότι είναι και για σας προτεραιότητα λόγω της ακρόασης που διοργάνωσε πέρσι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για τις νέες αυτές ψυχότροπες ουσίες και αυτό χάρη στον κύριο Σόνικ και την κυρία Ντονέσκου. Χάρη σε αυτού ε, διοργανώθηκε αυτή η άκρο επιτυχή ακρόαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται λοιπόν να παρουσιάσει αρχέ του 2013, του πρώτου μήνε του έτου αυτού, ε, πιο ισχυρέ προτάσει για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι νέε ψυχοτρόπε ουσίε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, πιο αναλογικά, πιο βιώσιμα. Ε, Στόχο είναι η βελτίωση τη ανταλλαγή των πληροφοριών και να γίνει αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά αυτέ τι ουσίε που δημιουργούν προβλήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και να αποσυρθούν γρήγορα από την αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέε ψυχοτρόπε ουσίε οι οποίε δημιουργούν προβλήματα κοινωνικά, προβλήματα υγείας, προβλήματα ασφάλειας. Και οι εναπομένουσε δύο νομοθετικέ προτάσει που ανακοινώσαμε για τα δικήματα όσον αφορά το εμπόριο ναρκωτικών και σχετικέ κυρώσει και το ευρύτερο πλαίσιο αναθεώρηση τη οδηγία για το ξέπλυμα πρόβλημικου χρήματο και αυτά θα παρουσιαστούν το 2013. Κυρίε και κύριοι, είναι πολύ σημαντική η νομοθεσία καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των ανταποκρίσεων, των αντιδράσεων για την αντιμετώπιση και της προσφοράς και της ζήτησης των ναρκωτικών. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας πολιτικής με τα ναρκωτικά είναι ο στόχος και αυτό είναι κάτι που το έχουμε εκφράσει μέσω πολλών στρατηγικών και σχεδίων δράση για τα ναρκωτικά. Είναι κάτι που το επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αναπτύξει ελάχιστε προδιαγραφέ ποιοτικέ για τη μείωση τη ζήτηση των ναρκωτικών, να βελτιωθεί η ποιότητα τη πρόληψη χρήση ναρκωτικών, θεραπεία και των υπηρεσιών κατά πολέμηση των συνέπειων ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με το Παρατηρητήριο για Ναρκωτικά Τοξικομανία που αναπτύσσει βασικού δείκτε για την για παραγωγή των ναρκωτικών, προμήθεια ναρκωτικών, την προσφορά ναρκωτικών αντιμετωπίσει τα προβλήματα τη αγορά ναρκωτικών, των εγκλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και να μειωθεί η προσφορά. Ο Βόλφκαν και εγώ στη Λισαβόνα πήγαν την περασμένη εβδομάδα και κάναμε τι πρώτε ομιλίε σε μια διάσκεψη Λισαβόνα. Είχαν έρθει περίπου 200 εμπειρογνώμονε για το θέμα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουν μια τεχνική συμφωνία όσον αφορά ε, δείκτες για την προσφορά ναρκωτικών και ετοιμάζουμε οδικό χάρτη για τους δείκτες αυτούς, για την προσφορά ναρκωτικών πριν κλείσω κυρίε και κύριοι να πω μερικά λόγια για τις ε, διεθνείς σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται στο διεθνές προσκήνιο όσον αφορά τη συζήτηση για τα ναρκωτικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδοθεί σε άκρο δραστήριο ε, διάλογο με χώρες παραγωγής ναρκωτικών ή χώρες διέλευσης ναρκωτικών καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διεξάγει πολιτικό διάλογο με αυτές τις χώρες, τους δίνει τεχνική και οικονομική βοήθεια και στήριξη Της βοηθά να δημιουργήσουν ε, δυναμικό για την αντιμετώπιση του εμπορίου ναρκωτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει εντατικότατο διάλογο με βασικούς εταίρους στην πολιτική των ναρκωτικών, παραδείγματος χάρη της ΗΠΑ Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ηγείται της ε, χρηματοδότησης προγραμμάτων για τα πολέμηση των παρανομενών ναρκωτικών. Το 2005 έχει και πέρα έχει δώσει 312 έχει εφαρμόσει προγράμματα αξίας 312 εκατομμυρίων ευρώ που βοήθησαν να δημιουργηθεί δυναμικό, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ναρκωτικών με πιο βιώσιμο τρόπο σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει επίσης πολυάριθμα προγράμματα για τα ναρκωτικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω χρηματοστικών προγραμμάτων, κυρίως ε, για την πρόληψη των ναρκωτικών και για την ενημέρωση των ναρκωτικά, το πρόγραμμα για την καταπολέμηση εγκληματικότητα και το πρόγραμμα για την υγεία το πρόγραμμα για την ενημέρωση για τα ναρκωτικά ήταν επιτυχέστατο και ήταν η ιδέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημιουργήθηκε χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2007 και μετά χρηματοδότησε πολυάριθμα προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτών πρόληψης και ενημέρωσης για τα παράνομα ναρκωτικά και ελπίζουμε ότι εν ώψη των νέων δημοσιονομικών προπτικών θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για να αντιμετωπιστεί και η ζήτηση ε, και η προσφορά ναρκωτικών και να γίνει ο αναγκαίος συντονισμός μεταξύ των δύο πτυχών. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Γιάκο Μπορατίνσκι από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών θέματα εσωτερικών, ο οποίος θα προσθέσει πληροφορίες σχετικά με προγράμματα και εξελίξει όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα, την πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο στην Επιτροπή για να συμπληρώσω την παρουσίαση που μας έκανε η Ντάνα. Όντως, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της συνολικής μας προσέγγισης ε, για το οργανωμένο έγκλημα και με τη νέα στρατηγική εσωτερική ασφάλεια που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θεωρήσαμε ότι η εξάρθρωση των διεθνών ε, κυκλωμάτων είναι βασικό μα στόχο και προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, θα ήθελα να τονίσω διάφορα σημεία. Καταρχήν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό το επιτυχάνουμε με τα ευρωπαϊκά συστήματα εποπτείας των εξωτερικών συνόρων. Έτσι εντομετωπίζουμε μικρά σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα που χρησιμοποιούνται για το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών. Στα εξωτερικά σύνορα επίση είναι σημαντικό να έχουμε μια κοινή ανάλυση και συνεργασία μεταξύ τη αστυνομία, των ε, σύνοροφυλάκων και των τελωνίων. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους ε, που ε, προκαλεί το οργανωμένο έγκλημα και ιδιαίτερα το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Έτσι, ετοιμάζουμε ε, την τέταρτη οδηγία για την ομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε το πακέτο της ε, Επιτροπή Μάστρομ που περιλαμβάνει την πάταξη της διαφθοράς, την εξάρθρωση τη σκιώδη οικονομία. Μερικές φορές οι λαθρέμποροι ναρκωτικών δωροδοκούν αξιωματούχου προκειμένου να διευκολύνουν την ε, είσοδο των ναρκωτικών στην ευρωπαϊκή αγορά και τώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την οδηγία περί κατάσχεσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος κεντρώνοντας την προσοχή μας ε, στο πιο σημαντικό θέμα που είναι τα κέρδη από τα ναρκωτικά. Το θέμα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών ε, ξέρετε ότι είναι η πιο επικερδής ε, εγκληματική δραστηριότητα του παρανόμου εγκλήματος και σίγουρα είναι σημαντική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθηση Ναρκωτικών και Τοξικομανία θα συνεργαστεί με τη Europol προκειμένου να καταρτιστεί νέα έκθεση, νέου είδου έκθεση για την αγορά των ναρκωτικών που θα δημοσιευθεί επίσημα στι αρχέ του επόμενου έτου. Στην έκθεση αυτή θα περιληφθούν σημαντικά επιστημονικά πορίσματα και η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθηση Ναρκωτικών σε συνδυασμό με ε, κάποιες ε, γνώσεις ε, για το οργανωμένο έγκλημα και θέματα πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα που έχει συγκεντρώσει η Europol. Μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις για παράδειγμα τον Ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος. Στα πλαίσια τη ε, στρατηγική εσωτερική ασφάλεια, τα κράτη-μέλη με την αρρωγή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, εκπονούν κάποιε προτεραιότητες ό,τι αφορά τη συνεργασία των διοκτικών του αρχών. Και μάλιστα οι σημαντικέ προτεραιότητε είναι εξή και πολλέ αφορούν τα ναρκωτικά. Είναι πολύ συγκεκριμένε αυτέ οι προτεραιότητε. Στηρίζονται σε μία στρατηγική ανάλυση και συμφωνία των κρατών μελών για το που η διασυνοριακή συνεργασία επιφέρει προστιθέμενη αξία. Οι προτεραιότητες είναι εξή. Θέλουμε να αποδυναμώσουμε την δυνατότητα, την ικανότητα των κυκλωμάτων οργανωμένων εγκλήματος που εδράζουν στην Αφρική, στη Δυτική Αφρική και ε, εισάγουν κοκαίνη και άλλα ναρκωτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσης, στα Δυτικά Βαλκάνια, που είναι βασική ζώνη διέλευσης ε, για παράνομα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των ε, ναρκωτικών, με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να αποδυναμώσουμε και αυτό το ρόλο. Επίσης, να μειώσουμε την παραγωγή και διανομή συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος ε, να παρεμποδίσουμε το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ιδιαίτερα κοκαίνης, ηρωίνης, κανάβεως και φυσικά την παραποίηση προϊόντων όπως τα σιγαρέτα. Είναι σημαντικέ οι προσπάθειε των κρατών μελών με τη συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να επικεντρωθούμε σε κέρια σημεία του λαθρεμπορίου ναρκωτικών που επηρεάζουν φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαιρόμαστε για την ευκαιρία που έχουμε να συγχαρούμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθηση Ναρκωτικών και τη Τοξικομανία για την παρουσίαση τη Γενική Έκθεση που θα ακούσουμε εντό ολίγου. Ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσω το λόγο στον κύριο Γκέτ, που είναι ο Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθηση Ναρκωτικών και Τοξικομανία. Θα μα παρουσιάσει τη Γενική Έκθεση του 2012. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να παρουσιάσω τα τελευταία ευρήματα του κέντρου σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών στην Ευρώπη. εκλήθη να παρουσιάσω και καινούρια στοιχεία για την τριετή στρατηγική μας ε, μέχρι το 2015. Η Ντάνα ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση των ναρκωτικών παραμένει μεγάλη πολιτική πρόκληση και η χρήση παράνομων ουσιών συνεχίζει να υπονομεύει τη δημόσια υγεία βλάπτοντας άτομα αλλά και οικογένειες και κοινότητες ολόκληρες και πολύ συχνά η χρήση και πώληση των ναρκωτικών ε, δημιουργεί παρεπόμενα προβλήματα. Πολλές προκλήσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε μια ρευστή αγορά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά συνθετικά φάρμακα και αυτά που επηρεάζουν τη διάθεση. Ε, υπάρχουν προκλήσεις, αλλά ε, είναι και ενθαρρυντικά τα νέα. <clears throat> Για ηρωίνη, κοκαίνη, κάναβη, Πολλές ε, χώρες ε, αναφέρουν μειούμενα επίπεδα κατανάλωσης. Ας δούμε τα οπιοειδή και την ε, ηρωίνη. Από τη δεκαετία του 70 η ηρωίνη ήταν το βασικό πρόβλημα στα μεταξύ των ναρκωτικών και θα έπρεπε να στις αρχές της δεκαετίας του 90. Γι' αυτό μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε το κέντρο μετά από μια πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου τότε του, του οι 1,4 εκατομμύρια χρήστες οπιοειδών ε, υπάρχουν, ε, δηλαδή ένας στους 250 ενήλικες. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η πολιτική ναρκωτικών επικεντρώθηκε στο να αντιδράσει αποτελεσματικά στα προβλήματα λόγω ηρωίνης και δημιουργήθηκαν μέτρα για να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα ε, των ε, ε, θανάτων, τη διάδοση του HIV και του ιού της υπατήτηδας και της κοινωνικής ζημίας που προκαλείται. Η ανάλυση μας δείχνει ότι μπορεί τώρα να μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου η χρήση ηρωίνης, ιδιαίτερα σε ενέσιμη μορφή, μπορεί να μειωθεί. Ε, μειώνονται οι νέοι χρήστες, αυτό είναι ένα, μια, μια ένδειξη. Ε, επίσης ε, μειώνονται αυτοί που κάνουν θεραπεία ε, και αυτό είναι μια άλλη ένδειξη. Υπάρχουν και δείκτες της αγοράς που υποδηλώνουν ότι η ηρωίνη είναι λιγότερο διαθέσιμη στην Ευρώπη. Τα τελευταία στοιχεία για την κατάσχεση και τα δικήματα δείχνουν αύξηση για διάφορους λόγους όμως. Στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ε, υπάρχει μια πρόσφατη έλλειψη ε, λόγω των επιτυχιών των διοκτικών αρχών και στην Εστονία και τη Φιλανδία η ηρωίνη αντικαταστάθηκε από συνθετικά οπιοειδή όπως φεντανίλ ή πουπρενοφίν. Ε, το, σήμερα ε, ε, βλέπουμε το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμων προσπαθειών μείωσης της προσφοράς και της ζήτησης. Επηρεάστηκε και ε, υπήρχαν μέτρα και στις οδούς διάθεσης της ε, ε, ηρωίνης αλλά και βελτιώθηκε η θεραπεία η οποία μείωσε τη χρήση της ηρωίνης. Σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις, πέρσι 1,1 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πήραν θεραπεία για τα ναρκωτικά και οι περισσότεροι πήραν υποκατάστατη θεραπεία. Περισσότεροι από τους μισούς ε, χρήστες του οπιοειδών είχαν πρόσβαση σε θεραπεία υποκατάστασης. Αλλά σε πολλές χώρες ακόμη ε, είναι ελλειπής η κάλυψη, ελλειπής οι ευκαιρίες. Τα σήματα επίσης μειώνονται. Ε, είναι, εξακολουθεί να είναι πρόκληση αυτή στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Υπήρχαμε έκρηξη του ιού του HIV, Πρέπει λοιπόν ε, να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα αυτό ε, μέσα από μέτρα και υπηρεσίες πρόληψης ε, από τη μόλυνση στο, από τον HIV. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Πολλοί τακτικοί χρήστες οπιοειδών πηγαίνουν για καιρό στη φυλακή. άλλοι έχουν καταστρεπτική συμπεριφορά. Ε, ε, το πρόβλημα οξύνεται ε, μετά την αποφυλάκηση και γι' αυτό θα πρέπει τότε να αντιδράσουμε και να παρέχουμε φροντίδα και στοχευμένα μέτρα για την αποκατάσταση της υγείας τους. Επίσης, αυξάνεται η χρήση των διεγερτικών. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλά χάπια, ε, επίσης κοκαίνη, αμφεταμίνη, έκσταση συνεχίζουν να παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο, αλλά σε, σε κάποιες χώρες βλέπουμε και καθενώνες μεθοτών MTPV, τα οποία προστίθενται στην αγορά των διαγερτικών. Η κοκαίνη όμως ε, είναι το δεύτερο ε, παράνομο φάρμακο μετά την κάναβη και περίπου 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν καταναλώσει το, την περασμένο χρόνο κοκαίνη. Όμως ε, δεν έχει τόσο το υψηλό στάτους που είχε παλιά και και σε κάποιες χώρες όπου η κατανάλωση είναι υψηλή, οι δείκτες δείχνουν ότι η χρήση φαίνεται ότι κορυφώθηκε και τώρα ακολουθεί καθοδική τάση. Για διάφορους λόγους. Η χαμηλή καθαρότητα κοκαίνη μπορεί να οδηγήσει στο πέρασμα σε άλλα διαγερτικά και οι δυνητικοί χρήστε μπορεί τώρα να γνωρίζουν τι αρνητικέ ε, ε, τις της περισσότερο. Ε, υπολογίζομαι ότι πέρσι 2 εκατομμύρια πήραν έκσταση, Ευρωπαίοι, και η αγορά του έκσταση πέρασε κάποιο μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια. Πρώτον, είδαμε σημαντική μείωση στα επίπεδα του MDNA, ε, MDMA ε, ε, στην έκσταση με ουσίες όπως BCP και μπεθατών στο έκσταση. Τώρα η αγορά του έκσταση φαίνεται ότι ε, έχει ανανύψει από την έλλειψη του MDNA και τώρα ε, υπάρχουν πάλι χάπια σε κάποιες χώρες που καταναλώνονται. Όμως ε, θα είναι το 100 ετών το υδραστική για το έκσταση, η οποία τότε ήταν ένα φάρμακο για να καταστήλει την όρεξη. Η αμφεταμίνη εξακολουθείται να χρησιμοποιείται στην Βόρεια Κεντρική Ανατολική Ευρώπη ε, περίπου 2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρησιμοποίησαν πέρσι αμφεταμίνες. Με η χρήση ε, των αμφεταμίνης σταθεροποιήθηκε για κάποια χρόνια. Τώρα όμως υπάρχουν ανησυχητικά δεδομένα για την μεθαμφεταμίνη. Στην Τσεχία και την Σλοβακία η μεθαμφεταμίνη ε, χρησιμοποιείται ε, αλλού είναι σπάνια. Από τη Βόρεια Ευρώπη επίσης, από την Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία, Γερμανία, ιδιαίτερα την Βαβαρία και τη Σαξονία, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η μεθαμφεταμίνη ε, ανεβαίνει. Ε, επίσης ε, ε αυξάνεται η χρήση διαγερτικών γενικότερα. Πριν από 10 μέρες είχαμε μία αξιολόγηση κινδύνου για τη μεθαμφεταμίνη στην ε, Λισαβόνα με, από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του κέντρου μας και διάφορες ε, υπηρεσίες και εμπλεκόμενα ε, μέρη. Κάναμε ομαδοποίηση θανάτων μιας μορφής αμφεταμίνης του MFTA που κατασκευάζεται σε κρυφά μυστικά εργαστήρια και ακολουθούνται ε, μυστικές οδοί ε, απόκτησης αμφεταμίνης για την παραγωγή. Ας δούμε τώρα τις ε, νέες ε, ψυχοτρόπες ουσίες. 49 νέες ουσίες ε, κοινοποιήθηκαν στο σύστημα πρόορις, ε, έγκαιρου συναγερμού στην Ευρώπη. Το 2012 ήδη ξεπέρασαν ε, το προηγούμενο ρεκόρ τους. 16 νέα μόρια επίσης για πρώτη φορά πρόσφατα ε, κοινοποιήθηκαν στο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης το 2012. Τα καναβοειδή και τα ε, ε, είναι ε, επίσης σε ανωδική πορεία. Σήμερα η αγορά ε, νέων φαρμάκων για λόγους αναψυχής αυξάνεται. Ε, σε εποχές μείωσης ε, έλλειψης της ηρωίνης τώρα κάνουν ένεση μεθοτρών ή MTPV, δηλαδή καθενοειδή. Σε κάποιες ομάδες νέων ανθρώπων είδαμε μεγάλη αύξηση στη χρήση νέων φαρμάκων και φαίνεται ότι το πρόβλημα οξύνεται διεθνώς. Ε, αυτές οι ουσίες ε, δεν ξέρω, ε, δημιουργούν μεγάλες απειλές στην πολιτική μας. Στηρίζομαι τους πολιτικούς καθώς προσπαθούν να αντιδράσουν αποτελεσματικά και η νομική βάση του συστήματος ε, Προειδοποίηση ε, και ανάλυση κινδύνου ανανεώνεται. Η Ντάνα το ανέφερε αυτό. Πρέπει να βελτιώσουμε την, ε, τις ε, ε, ε, ιατροδικαστικές μας δυνατότητες και σε σχέση με τις νέες ψυχοτρόπες ψυχοδραστικές ουσίες. Θα πρέπει να καταλάβουμε την επίδραση αυτών των φαρμάκων στην υγεία για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Τα τελευταία χρόνια οι παλιές νέες ε, ουσίες ε, ε, εγκαταστάθηκαν στην αγορά. Μιλάω για φάρμακα όπως CHB, κεταμίν και νιουμεθοτρόν. Ο συνολικός αριθμός των χρηστών παραμένει χαμηλός και έτσι ξεγλιστρούν από το ραντάρ παρακολούθησης. Υψηλά επίπεδα κατανάλωσης εντοπίστηκαν σε ορισμένες ομάδες νέων. Επίσης είδαμε και σοβαρά οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας σε σχέση με τη χρήση αυτών των ουσιών. Αυτές οι εξελίξεις μας θυμίζουν ότι το, πολλές φορές το τωρινό μα όραμα είναι περιορισμένο και δεν μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε και να αντιοπίσουμε νέες απειλές. Ας δούμε τώρα την κατάσταση στην κάναβη. Η τελευταία ανάλυση μας στην αγορά της κάναβης δείχνει ότι η παραγωγή στα σύνορα της Ευρώπης αντικαθιστά την εισαγόμενη κάναβη. Ε, η τοπική αγορά κανάβεως ε, κυμαίνεται από μικρούς καλλιεργητές ε, για προσωπική χρήση μέχρι μεγάλες φυτίες που χρησιμοποιούν εκλεπτισμένες τεχνικές. Η κάναβη συνεχίζει να είναι το πιο σύνηθες παράνομο ναρκωτικό. 23 εκατομμύρια ήταν οι χρήστες πέρσι, όπως εκτιμάται. Δηλαδή ένας στους 15 ενήλικες. Μεταξύ αυτών 3 εκατομμύρια ενήλικες που χρησιμοποιούν κάναβη σε καθημερινή, σχεδόν καθημερινή ε, βάση. Αυτό είναι σημαντικό. Τα προβλήματα της, ε, σχετικά με την κάναβη ε, δεν κατανοούνται πολλές φορές, ε, αλλά πολλές φορές συσχετίζονται με την εντατική και μακροχρόνια χρήση του φαρμάκου, του ναρκωτικού. Η φυτική κάναβης μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε πιο ισχυρές μορφές του φαρμάκου και στην Ευρώπη υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ατόμων που κάνουν θεραπεία για τα προβλήματα από την κάναβη. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση αυτή, η καινούρια μας έκθεση, ε, δείχνει την σύνθετη και διαφοροποιημένη φύση του προβλήματος των ναρκωτικών. Ε, πολλά από αυτά που έχουμε είναι και καλές, καλά νέα. Ε, πολλές φορές ακούγονται και απεσιόδοξε φωνές που αμφισβητούν τις επιτυχίες των προσπαθειών μας. Νομίζω ότι αν δούμε προσεκτικά τα στοιχεία βλέπουμε εύκολα ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση που αναγνωρίζει ότι προσφορά και ζήτηση έχουν ίση σημασία που αναγνωρίζει την αξία της επιστημονικής και τεκμηριωμένης προσέγγισης που είναι ρεαλιστική, που αξιολογεί τις δράσεις και πάνω απ' όλα που αναγνωρίζει την ανάγκη να ε, ε, προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμους στόχους, αυτή η προσέγγιση κάνει διαφορά. Δεν μπορώ βέβαια να παραλείψω να πω δύο λόγια προειδοποίησης αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις έχουν να κάνουν ε, επιλογές δύσκολες, ε, οι προτεραιότητες είναι δύσκολες. Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να γίνουν σοφές επενδύσεις ε, στα παράνομα ναρκωτικά. Επενδύσεις πάνω στη σωστή κατανόηση του προβλήματος και των μέτρων που θα δώσουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Η πρόοδος που παρατηρήσαμε μπορεί να αντιστραφεί αν οι επενδύσεις σταματήσουν ενώ ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικέ. Όπω είπαμε σήμερα, η αγορά των ναρκωτικών σήμερα είναι δυναμική, καινοτόμο και γρήγορα ανταποκρίνεται σε προκλήσει. Ε, για να ανταποκριθούμε, συνεργαζόμαστε με τη Europol σε μια στρατηγική ανάλυση σε βάθος, όπως ανέφερε και η Ντάνα προηγουμένως. Και τον Ιανουάριο του 2013 θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά μας. Ε, η έκθεση στις 15 Νοεμβρίου κοινοποιήθηκε και παρουσιάστηκε μαζί με την Επίτροπο Μάλμστρομ ε, στην έδρα μας στη Λισαβόνα ε, με 45 δημοσιογράφους παρόντες που ήρθαν ως ειδικά για αυτή την εκδήλωση στην Λισαβόνα αλλά υπάρχουν και δημοσιογράφοι διεθνούς ρεπορτάζ που είναι στη Λισαβόνα μόνιμα. Επίσης έγιναν, παρουσιάστηκε το θέμα και σε εθνικό επίπεδο, σε άλλες χώρες. Η τελευταία παρουσίαση θα γίνει 11-12 Δεκεμβρίου στην Πορτογαλία σε μια ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας του ε, Πορτογαλικού Κοινοβουλίου. Μετά από μια εβδομάδα κάλυψης ε, από τα ΜΜΕ, ε, είδαμε και ε, ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν ε, πάρα, πολλά, πάρα πολλές καλύψεις. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε 1.500 μέχρι 2.000 αναφορές από τα ΜΜΕ όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Και στην Νορβηγία, Κροατία, Τουρκία, τρει χώρε που συνεργάζονται πολύ στενά έχουν μεγάλη κάλυψη. Τη μεγαλύτερη κάλυψη την είχαμε στη Γερμανία, Ισπανία και Γαλλία. Διεθνώ ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία έχουμε τη μεγαλύτερη κάλυψη και είχαμε αύξηση στο Καναδά, το Μεξικό, την Ταϊβάν, τη Βενεζουέλα, τις Αραβικές χώρες και την Ουκρανία. Παραδόξως ε, δεν είδαμε ανάδραση από την Κίνα και την Νότιο Κορέα όπου πάντοτε ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλές αναφορές. Θα περιμένουμε λίγο ακόμη. Η έκθεση ανεβάστηκε πάνω από 18.000 ε, φορές ε, και στα αγγλικά, ισπανικά. Υπάρχει, είναι διαθέσιμη άλλωστε σε 22 γλώσσες. Ε, από τη 22.000 το 60% είναι κατανεμημένο και είδαμε και αναφορές πριν από το λανσάρισμα. Ας περάσουμε τώρα στο νέο ευρωπαϊκό, στο νέο στρατηγική του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης 2013-2016 έχουμε το τρίτο πρόγραμμα εργασίας μετά τον κανονισμό αναδιατύπωσης που τέθηκε σε ισχύ το 2007 και που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώθηκε και με τη συνεργασία της Επιτροπής σας. Το πρόγραμμα εργασίας αυτό στηρίζεται στα θεμέλια ε, του έργου του παρατηρητηρίου και θέλει, θέλουμε να εξασφαλίσουμε την παρακολούθηση της σύγχρονης κατάστασης ό,τι αφορά τα ναρκωτικά. Κατά την κατάρτιση του φετινού προγράμματο ε, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τους εξωτερικούς παράγοντες και τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το έργο μας την επόμενη τριετία. Έχουμε φυσικά το θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, οι περικοπές των πόρων στα κράτη-μέλη, προκλήσεις ε, και νέες απαιτήσεις από τους οργανισμούς. Και φυσικά Δυστυχώς ε, υπάρχουν πολλές πολλά αιτήματα για χρηματοδότηση, αλλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά. Και φυσικά θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους, ε, ώστε να ληφθούν υπόψη οι στάσεις τους και οι ανάγκες τους. Και τελευταίες ε, διαδικασίες διαβούλευσης έγιναν με τα κράτη-μέλη, με τα, με θεσμικά όργανα, με την Επιστημονική Επιτροπή, με τα γραφεία επαφής, με άλλους οργανισμούς δικαιοσύνης εσωτερικών, φαρμάκων και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παρακολούθηση των Νόσων με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και φυσικά και με το κοινό. Λάβαμε υπόψη στις διαβουλεύσεις αυτές ε, τις συστάσεις και ε, της τρίτης εξωτερικής αξιολόγησης του κέντρου μας που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ παραλίλου με τις δικές μας διαδικασίες προγραμματισμού. Και η αποστολή μας για την επόμενη τριετία είναι να προβούμε σε μια σφαιρική ανάλυση της κατάστασης των ναρκωτικών ε, περνώντας ε, σε ένα ε, μετατρέποντας το κέντρο μας σε ένα πραγματικό κέντρο ανάλυσης. Έχουμε βασικές αρχές και προτεραιότητες. Για παράδειγμα, θέλουμε να προβούμε σε μια επίκαιρη και έγκαιρη ανάλυση της κατάστασης των ναρκωτικών, να αξιοποιήσουμε τις δραστηριότητες και τις απενδύσεις στο έπακρο και η τρίτη μας αρχή και προτεραιότητα είναι καλή επικοινωνία και μια προσέγγιση που θα προσανατολίσει τις ανάγκες των χρηστών των πελατών μας. Έχουμε επίσης πέντε θεματικές προτεραιότητες. Θα πρέπει να αντιληφθούμε το πρόβλημα, να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις καλύτερες πρακτικές αντίδρασης, νέες στάσεις, εξελίξεις, υποστήριξη των πολιτικών και πέμπτον ε, αναβάθμιση το, της ενημέρωσης για την προσφορά και τις αγορές. Τώρα, πώς θα μεταφέρουμε μετατρέψουμε σε έμπρακτα αποτελέσματα αυτό το στρατηγικό μας όραμα. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα για το νέο μας πρόγραμμα εργασιών. Καταρχήν, το πρώτο παράδειγμα αφορά την ετήσια μας έκθεση. Η έκθεση αυτή με τη μορφή που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι η τελευταία. Από το 2013 και μετά θα δίνουμε στο κρατήριό μας και στους ενδιαφερόμενους ε, μία νέα έκθεση που θα ακολουθεί ένα τελείως διαφορετικό κόνσεπτ και αντίληψη. θα είναι πολύ πιο επίκαιρη, θα ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογίες, ε, στις ανάγκες του ίντερνετ και των κοινωνικών μέσων, αλλά και στο γεγονός ότι έχουμε λιγότερους πόρους. Θα έχουμε μια πολύ πιο εστιασμένη ανάλυση της κατάστασης των εργατικών στην Ευρώπη, θα έχουμε μια έκθεση πολύ πιο σύντομη, βέβαια θα μεταφράζεται και πάλι στις 22 γλώσσες και θα δίνεται ένα πεντάμινο νωρίτερα. Οπότε την επόμενη φορά θα με δείτε πολύ πιο νωρίς από αυτή τη φορά. Η ετήσια έκθεση δεν είναι ένα απλό προϊόν. Είναι ένα τμήμα ενός ευρύτερου πακέτου. Και τα περισσότερα τμήματα αυτού του πακέτου χορηγούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, με ηλεκτρονικό υπόθεμα. Έτσι θα δώσουμε μια πιο ξυδερκή ανάλυση της, κατα... της... του έργου μας, μια πολύ σύγχρονη και επίκαιρη πολύ πιο σύγχρονη και φυσικά θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και τον τίτλο. Οι περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται online περισσότερο, μέσω του διαδικτύου και όχι ε, με γραπτή μορφή. Και θα επικεντρωθούμε σε θεματικές ενότητες. Υπάρχει φυσικά και το στατιστικό σκέλος που ήδη υπάρχει στο ίντερνετ, ε, ένα σύνολο πινάκων και στατιστικών στοιχείων που θα είναι πιο διαδραστικό, θα έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες για τα προφίλ των χωρών, οπότε ο καθένας θα μπορεί να, δει, να, διαπιστώνει τι θέση έχει η χώρα του στο, στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η ενίσχυση του συστήματος παρακολούθησης μας και του αναλυτικού μας έργου πέραν της ενίσχυσης του συστήματος παρακολούθησης ε, για το σκέλος της ζήτησης, γιατί πολύ συχνά αναφερθήκαμε στους ε, πέντε βασικούς μας δείκτες ε, στον τομέα της επιδημιολογίας. Θα έχουμε τώρα νέους δείκτες για την προσπάθεια μείωσης της ζήτησης, για τα χαρακτηριστικά των αγορών ναρκωτικών και πριν από λίγο η Ντάνα μας μίλησε για τη δεύτερη διάσκεψη για τους δείκτες ό,τι αφορά την ε, προσφορά των ε, ναρκωτικών. Επίσης, ό,τι αφορά το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ανάλυση των κινδύνων, των μηχανισμών ανάλυσης κινδύνων. Θα οργανώσουμε ε, την σημαντική μελέτη για τα δημοτικά σχολεία, την ΕΣΠΑΤ, που υπάρχει από το 1993. Μέχρι στιγμής την διοργάνωνε η Σουηδία, θα το αναλάβουμε πλέον εμείς. Και το τελευταίο παράδειγμα, πριν ολοκληρώσω, είναι ότι θα ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε η διαδικασία και η πολιτική μας θα γίνει πιο αποτελεσματική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συνδράμουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη νέα στρατηγική της για τα ναρκωτικά που σας παρουσίασε πριν από λίγο η Ντάνα και θα συνεχίσουμε φυσικά να στηρίζουμε και τα μεμονωμένα κράτη-μέλη την προσπάθεια ανάλυσης των στρατηγικών τους, εφόσον φυσικά μας ζητηθεί μια τέτοια συνδρομή, και θα συνεχίσουμε ε, να εφαρμόζουμε τις δραστηριότητες μας ε, που μας έχουν ανατεθεί και στη συνεργασία με τη Γεροπόλ και στα πλαίσια του σχεδίου δράσης COSI. Αυτά προς το παρόν. Μπορώ να ολοκληρώσω εδώ την παρουσίασή μου και σίγουρα με το νέο πολιτέ πρόγραμμα θα συμβάλλουμε στη χορήγηση καλύτερη ε, πληροφορία και ανάλυση ώστε να ανταποκριθούμε καλύτερα στα προβλήματα ναρκωτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ε, λάβουμε και τις αποφάσεις για την ε, οριστικοποίηση του πρώτου έτους από το τριετέ πρόγραμμα εργασιών. Ευχαριστώ κύριε Γκέτς. Έχουμε να μιλήσουν ο κύριο Γιακολίνο, κυρία Ζίπελ και η κυρία Λόπες Ο Γιακολίνο. Θα είστε σύντομος παρακαλώ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε, ακούσαμε e τις πολύ εμπεριστατωμένες αυτές παρουσιάσεις. Πρώτα από την κυρία Ντάνα Σπίνα που την ευχαριστώ και τον διευθυντή Wolfgang Γκέτς Αναμφισβήτητα το 2012 όπως λέει, ε, συμπίπτει η ετήσια έκθεση με την ολοκλήρωση του προγράμματος για την στρατηγική καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένη αξιολόγηση της επταετίας των δραστηριοτήτων. Μια στρατηγική που ουσιαστικά λειτουργήσε με πόρους που δεν ανταποκρινόταν πάντα στους στόχους, βλέποντας ότι αυξάνεται η αγορά, το μέγιστο της αγοράς, μπαίνουν νέα ναρκωτικά, συνθετικά, που μπαίνουν στην αγορά από τη μέρα στην άλλη. Έχουμε φτάσει στα 60 του 2012. Από 40 σε 60 ανεβήκα σε ένα χρόνο. Και υπάρχουν και διαφορετικές νομοθεσίες σε κάθε χώρα. Κάθε κράτος ακολουθεί διαφορετική πολιτική αντικαταπολέμηση ναρκωτικών, προσοχή που δίνει στους νέους, καταπολέμηση της προσφοράς κλπ. Θα πάω κατευθείαν στο θέμα το οποίο θέλω να θίξω. αυτό που σχετίζεται με την φυσική και ψυχολογική υγεία εκείνων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βόλφκαν Γκότς αναφέρθηκε στους νέους. Εγώ θα έλεγα ότι το νέο πρόγραμμα, θέλω να αναφερθώ στο νέο πρόγραμμα 2013-2015. Ποια θα είναι η δετομεϊκή προσέγγιση. Για πρώτη φορά στην έκθεση γίνεται ρητή αναφορά στις συμπεριφορές, στην συμπεριφορά, στην εξάρτηση, στις συμπεριφορές εξάρτησης και πώς πρέπει να ακολουθηθεί η διατομική προσέγγιση όσον αφορά την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Ποια θα είναι αυτή η διατομική προσέγγιση για να λάβουμε υπόψη και άλλες τοξικομανίες πέραν από αυτέ που συνδέονται με τις ψυχοτροπικές ουσίες. Και ποια θα είναι η προσέγγιση όσον αφορά την τοξικομανία και των φυλακισμένων. Ένα τρίτο του πληθυσμού των φυλακισμένων χρησιμοποιεί ε, τέτοιες ουσίες. Χρησιμοποιεί ναρκωτικά. Και πρέπει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να διαπιστωθεί ποια θα μπορεί να είναι η ενία αντιμετώπιση που θα μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόληψη όχι στα πλαίσια της δικαιοσύνης όπου προσπαθούμε να μειώσουμε παραγωγή και εισαγωγές ναρκωτικών, αλλά ε, σε σχέση με τα προβλήματα ομάδων του πληθυσμού, όπως ανέφερε και ο κύριος Γιακολίνο, και σε σχέση με τη δικτύωση. Η πρόληψη των ναρκωτικών ε, στρέφεται κυρίως στους νέους και πώς γίνεται η πρόληψη. Ενημερώνουμε και προειδοποιούμε για τις τρομακτικές συνέπειες ε, της ε, χρήσης. Επίσης πρόκειται για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αυτή είναι μια προσέγγιση που τη γνωρίζω από τη δεκαετία του 80 και πράγματι θα πρέπει να δούμε πώς οι διάφοροι τομείς των πολιτικών μας θα ε, διασυνδεθούν καλύτερα και για, καλύτερη, για μεγαλύτερη επιτυχία. Ε, επίσης υπάρχουν κάποια στοιχεία αν ομάδες του πληθυσμού στα νόμιμα και παράνομα ναρκωτικά ε, πλήττονται ιδιαίτερα από τη χρήση ούτως ώστε να είμαστε πιο στοχευμένοι στα μέτρα που θα λάβουμε. Γενικά η εντύπωσή μου είναι και θα ήθελα μια επιβεβαίωση ή διευκρίνηση ότι δεν χρειαζόμαστε καταρχήν συνεχώς καινούργια νομοθεσία, αλλά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας θα πρέπει να διασυνδέσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας για πιο ευέλικτη αντίδραση και νομίζω ότι και σε επίπεδο κρατών μελών ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερη ευαισθητοποίηση ε, και να δούμε τους διάφορους τομείς που κατά πρέπει να δούμε μαζί. Ευχαριστώ κυρία Λόπες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση για τους θανάτους από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Η έκθεση αναφέρει ότι στο 2009 είχαμε 7.600 κρούσματα υπερβολικής δόσης και οι μισές περιπτώσεις, τα μισά κρούσματα ήταν στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για το 2010 έχουμε 7.000 θανάτους. Είχαμε μείωση λοιπόν των μοιραίων περιστατικών. Επίσης, ε, για, τα καναβοειδή είχαμε τη, το 2010 τις περισσότερες περιπτώσεις ε, στην Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Κροατία, στις χώρες του Νότου. Δεν καταλαβαίνω πώς καταρτίζετε αυτούς τους χάρτες και πώς καταλήγετε σε αυτά τα στοιχεία. Έχω την αίσθηση ότι για τους θανάτους από υπερβολική δόση ναρκωτικών θα έπρεπε να αφιερώσουμε περισσότερη προσοχή στην έκθεση. γιατί δεν γίνεται μία ανάλυση των τάσεων. Από το 2010 και μετά δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε τα επίκαιρα στοιχεία, δεν ξέρουμε πώς εξελίχθηκαν οι συμπεριφορές στις διάφορες χώρες. Αναφέρονται κάποιοι πολύ γενικοί και όριστοι λόγοι. Έλλειψη θεραπείας, προβλήματα οικογενειακά. Σε ποιες χώρες δεν υπάρχει τέτοια θεραπεία ή δεν υπάρχει υποκατάστατη θεραπεία. Ε, οι πολυτοξικομανίες, ε, η παραντερολογική πολυτοξικομανιες η παρατερολογικη οδος θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν πραγματικά η φυλακή ε, ασκεί επιζήμια επίπτωση στην υγεία των τοξικομανών. Έχουμε στοιχεία για τοξικομανείς ε, που είναι φυλακισμένοι. Μας ενδιαφέρουν τέτοια στοιχεία, γιατί είναι συναφή τα στοιχεία αυτά με την πολιτική μας για την κατανάλωση των ναρκωτικών σε ποιε χώρες είναι αξιόπινη η κατανάλωση ναρκωτικών και σε ποιες όχι. Επίσης, να γίνει μια εκτίμηση των θανάτων από υπερβολική δόση. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, το στοιχείο αυτό για να δούμε τι πολιτική εφαρμόζει κάθε χώρα. Δυστυχώ μιλούν ταυτόχρονα η πρόεδρο και η κυρία Λόπες. Ναι. Διακόπτει η πρόεδρος την κυρία Λόπες. Η ναι. κυρία Ντάνα Σπίνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα απαντήσω συντομία στις τρει ε, ερωτήσει. και κατόπιν θα δώσω το λόγο στο Wolfgang που θα δώσει πιο ουσιαστικές ε, απαντήσεις από την ετήσια έκθεση. Απαντώντας στον κύριο Γιακολίνο, θα ήθελα να πω ότι όντως είναι πολύ εύστοχο αυτό το σχόλιο του ότι η τοξικομανία θα πρέπει να θεωρηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στο πλαίσιο των εθισμών. Γιατί πολλές φορές οι μηχανισμοί, οι νοητικοί μηχανισμοί για τους εθισμούς είναι παρόμοιοι. Η νέα στρατηγική των ναρκωτικών ε, τονίζει την σημασία ε, της ανάλυσης όχι μόνο των παράνομων ναρκωτικών αλλά και των νόμιμων ουσιών που χρησιμοποιούνται. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί είναι ένα μείζον ερευνητικό πρόγραμμα για τον εθισμό και τον τρόπο ζωής. Λέγεται Alice Rap και θα ολοκληρωθεί το 2016. Πρόκειται για ένα σχέδιο που χρηματοδοτείται με 10 εκατομμύρια ευρώ από το 7ο Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο. Και θα μας δώσει νέες στοιχείες για το σχετισμό των ε, εθισμών με νέες ε, ουσίες, αλλά και θα αναλύσει γενικώ τις εξαρτημένες συμπεριφορές. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο της κυρίας Ζίπελ για την πρόληψη, όντως η πρόληψη είναι τομέα που υπάγεται ε, κυρίως στις εθνικές αρμοδιότητες λόγω της αρχής επικουρικότητας. Η νέα στρατηγική των αρκετικών τονίζει την ανάγκη... Συγγνώμη που σας διακόπτω, λέει η Πρόεδρος. Καθίστε παρακαλώ, συνάδελφοι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες αν δεν ολοκληρώσουμε την προηγούμενη μας συζήτηση. Η νέα στρατηγική λοιπόν για τα ναρκωτικά τονίζει την σημασία της πρόληψης γιατί εκεί πραγματικά ξεκινά το, το πρόβλημα των ναρκωτικών. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε διάφορες πτυχές πρόληψης, ε, οικομενικής, εστιασμένης, περιβαλλοντικής πρόληψης και να αξιολογήσουμε και την αποτελεσματικότητα των ε, προγραμμάτων πρόληψης. ευχαριστώ και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κέτς. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, χρόνου φίδου. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα είμαι συντομότατος. Το πρώτο που έθεσε ο κύριος Γιακολίνο για άλλους για άλλες εξαρτήσεις και σχέση μεταξύ παρανόμων ουσιών και νομίμων είναι σημαντικό θέμα. Έχουμε δύο προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη στη Νότια Ευρώπη, Κέντρο και Νότια Ευρώπη, εστιάζονται οι προσπάθειες στον εθισμό και όχι στο κατά πόσο είναι παράνομες οι νόμιμες ουσίες. Ή αν ο εθισμός ε, είναι άλλο είδους εθισμός, όπως μπορεί να, το να στοιχηματίζει, να παίζει κανείς και δεν σχετίζεται με ουσίες στη Βόρεια Ευρώπη και στις χώρες γίνεται διάκριση και η εντολή του κέντρου παρατήρησης είναι, στις, ε, είναι περιορισμένη στις παράνομες ουσίες. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στον τομέα. Και για να κινηθούμε όλοι μαζί με τον ίδιο τρόπο στην Ευρώπη. Όσον αφορά την πρόληψη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας τομέας μείωση ζήτησης ναρκωτικών. το πάντα με πολιτική βούληση και όχι μέσω στοιχείων. Άλλαξε η προσέγγιση τελευταία χρόνια. Γίνεται καλύτερη εξολόγηση προγραμμάτων πρόληψης. Η προσέγγιση σήμερα είναι κάτι παλιό, θα λέει η κυρία Ζίπελ. Θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά και στους νέους αξίες και τρόπους συμπεριφοράς και αντίδρασης. Για να δείξουν ότι να αντέχουν την πίεση της ομάδας τους, ότι είναι, αυτός που τα αντέχει είναι δυνατός. Και μετά εστιάζονται επί των ομάδων. Κάτι που δεν είναι πολιτικό ορθό. Αυτό βλέπουμε να γίνεται σήμερα παρόλα αυτά. Και είναι επιτυχές να επικεντρώνουν οι προσπάθειες σε ευάλωτες ομάδες. Η κυρία Ρομέρο Λόπες αναφέρθηκε σε κάποια θέματα. Πολλά στοιχεία μας της εκθέσεως είναι του 2010. Είναι κάπως παλιά στοιχεία, αλλά είναι όλη η διαδικασία που αργεί, η μετάφραση κλπ. Γι' αυτό θέλουμε πιο γρήγορη διαδικασία τάξη εκθέσεων. Η επόμενη θα εκδοθεί τον Μάιο. Όσον αφορά τις πληροφορίες που λείπουν, η έκθεση είναι ένα μόνο κομμάτι ενός πακέτου και το πακέτο εκθέσεων συμπεριλαμβάνει και στατιστικά στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που δεν παρουσιάσαμε σήμερα και που δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Αυτό ήταν το σημαντικότερο που είχα να σας πω. Δημερός μας συνεχίσουμε όμως. Ήθελα να είμαι σύντομο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ κύριε Γκέτς. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, οι σκέψεις σας.

Okay. Colleagues, let's continue with the votes. Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες. We most probably will need voting cards. Θα χρειαστείτε τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Ελπίζω να τις έχετε όλες. Σημείο 14. Πρώτη απόφαση θα γίνει μια ψηφοφορία προσανατολισμού όσον αφορά προγράμματα ανταλλαγή και κατάρτισης για την προστασία του ευρώ κατά της ε, παραχάραξης. Η κυρία Μάκιντάρ είναι η συγγήτρια και θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Μάκιντάρ, είχε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Έκλεισε το μικρόφωνο τη κυρία Μάκιντάρ και δεν μπορούμε να ακούσουμε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο σύντομα σχόλια έχω. Πρώτον, Ευχαριστώ πολύ τον αποσιάζοντα πρόεδρο γιατί διευκρίνησε τη θέση για τις κατεξουσιοδότητες συμπράξεις. Ενημέρωσα δεόντως τους Σκιώδης και ελπίζω ότι θα τύχουμε υποστήριξης για τρεις σχετικές τροπολογίες 35, 15 και 1 που υποστηρίζουν την απόφαση του Κοινοβουλίου για τις κατεξουσιοδότης πράξεις. Άλλος τομέας στον οποίο υπήρξε κάποια διαφωνία ήταν η, τα ποσοστά συγχρηματοδοτήσεως. Ακολούθησα ρεαλιστική προσέγγιση. Θεώρησα ότι είναι σημαντικό το πρόγραμμα να συνεχιστεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, μία μειοψηφία στο ε, Σκηνοβούλιο, αναστέλουσα μια ψηφία και 15 προσπαθεί να διατηρήσει τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που υπάρχουν γιατί αν το υποστηρίξουμε αυτό πιστεύω θα σημειώσουμε πρόοδο και θα περάσει το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους στην υποστήριξή τους και που με βοήθησαν. Και θράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω τον Άλντο από τη Γραμματεία την καλή του δουλειά και να του ευχηθώ καλή τύχη στο μέλλον. Σας ευχαριστώ κυρία Μάκεντάιρ. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Τροπολογία 26, συγγνώμη. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική σι λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά πρέπει να γίνει έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 35 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Κυρία Ρόμαντσα, βάλατε την κάρτα σας, έτσι. 29 υπέρ, 19 κατά. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 Α, πάμε σε τελογικές σκέψεις. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ αψηφίστηκε με 35 και 15 πάμε λοιπόν στην τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 48 ψήφοι πέρα. Καμία αποχή. Δεν υπάρχει ψήφος εναντίον. Συγχαρητήρια λοιπόν, κυρία Μακεντάιρ. Πάμε στο άλλο σημείο, στο δεύτερο σημείο, στον κατάλογο ψηφοφοριών ψηφοφορία όσον αφορά την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει τι γενικέ διατάξει για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευση και τα εργαλεία για την οικονομική υποστήριξη, για την αστυνομική συνεργασία, για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματο και τη διαχείριση των κρίσεων. Η Εισηγητή είναι ο κύριο Φοντάνα. κυρία Σαρτζεντίνη. Δεν ακούγεται η κυρία Σαρτζεντίνη. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, η πράσινη θέλουν να αποσυρθούν τη συμβαστική τροπολογία 9 η τροπολογία της συναδέφα Τσέσκα Κέλλερ, η 133, αναφέρεται στη τροπολογία 9. Δεν θεωρούμε ότι συμφωνούμε με αυτή. Η συγγήτρια ποτέ δεν μας προσήγγισε, απλώς έβαλε το όνομά μας και θέλουμε να αποσυρθούμε από τη συμβαστική τροπολογία 9. Ευχαριστώ, ας ψηφίσουμε. Ξεκινάμε με την τροπολογία 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται τροπολογία 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60 είναι η γλωσσική φύσεως, δεν ψηφίζεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 και 18 της Επιτροπής Υπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 και 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Έλεγχος για τη συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 35 με 13 εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν αποχές. Πάμε στην 72 υπέρ κατά αποχές ορίστε δεν λειτουργήσε ούτε μία φορά η ηλεκτρονική μου κάρτα ψηφοφορίας το δήλωσα στη γραμματεία Αντικαθιστώ το Χουαν Φερνάντο Λόπε Αγγιλάρδα. Δυστυχώ ούτε μία φορά δεν κατάφερα να ψηφίσω με την ηλεκτρονική μου κάρτα. Δεν λειτουργήσε ούτε μία φορά. Προσπαθείτε να, προσπαθήστε να βρείτε μια άλλη, να βρείτε μια άλλη θέση. Τρει φορέ άλλαξα θέση. Ίσως έχετε πρόβλημα με την κάρτα σας εν τη αυτή περίπτωση. 48 ψήφισαν όμως. Πρέπει να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Και θα σας μετρήσουμε ξεχωριστά, λοιπόν. Τροπολογία 72 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Τροπολογία Έλεγχος λοιπόν για την τροπολογία 9, ηλεκτρονικός. Λειτουργεί το μηχάνημά σας τώρα. Ωραία. 33 υπέρ, 16 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Πάμε στην 76 υπέρ, κατά. Άλλη μια φορά. 76 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται διορθώνει πρόεδρος. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε για την τροπολογία 80 ηλεκτρονικός έλεγχος Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 17 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται λέει η Πρόεδρος. Τι είπα λέει η Πρόεδρος, συγγνώμη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, συγγνώμη λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές ξανά 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στην τροπολογία τροπολογία 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά έλεγχος έλεγχος για την τροπολογία 89 ξεκινάει η ψηφοφορία Τέλος. 21 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 88 υπέρ, κατά, αποχές Α, ήταν ταυτόσιμες. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 με προφορική τροπολογία και κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε στην τροπολογία 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 98 υπέρ, καταπίπτει, συγγνώμη, συγγνώμη, 99 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται, 22 της Επιτροπής υπέρ, Α, συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Πάμε στην 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 103 υπέρ, 102 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά α, δεν βλέπω 105 έλεγχος ξεκινά ο ηλεκτρονικός έλεγχος 19 υπέρ, 30 κατά, σαφώς απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 έχει ένα λάθος στο αγγλικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 καταπίπτει 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές σηκώνετε το χέρι σας παρακαλώ είναι πολύ δύσκολο να σας δω 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στην 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται εγκρίνεται εγκρίνεται έλεγχος για την 118 ηλεκτρονικός έλεγχος ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας 34 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 Έλεγχος για την 124. Ξεκινάει η ψηφοφορία. 124. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 125 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 και 24 υπολογισμών υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Πιθανότατα εγκρίνεται. Έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 21 ψήφοι κατά, 4 αποχές. Εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135 υπέρ, κατά, αποχές αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά Έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 142. Ξεκινάει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 23 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ κατά αποχές άλλη μια φορά 144 σηκώστε το χέρι παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά ξανά παρακαλώ σηκώστε το χέρι όλοι είναι πολύ δύσκολο 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, εγκρίνεται διορθώνει ο πρόεδρος, 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. 26 προπολογισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 προπολογισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 28 προπολογισμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 162 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 162, άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε συνάδελφε. Καλώς, πέρας ψηφοφορίας, 29 υπέρ, 19 κατά εγκρίνεται. 29 προπολογισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 170 ξεκινάει η ψηφοφορία Πέρα ψηφοφορία. 22 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. Προϋπολογισμού 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προϋπολογισμού 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, α, Πρέπει να γίνει έλεγχος για την 171. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται διορθώνει η πρόεδρος ζητώ συγγνώμη 187 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 187 άρχεται η ψηφοφορία Πέραση 27 υπέρ 24 ψήφοι κατά εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τρο... πάμε σε τελογικές σκέψεις σε αναφορές τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εγκρίνεται εγκρίνεται ζητώ συγγνώμη λέει ο πρόεδρος προπολογισμού 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προπολογισμό 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 καταπίπτει 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμόν 11 υπέρ, κατά, άλλη μια φορά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προϋπολογισμόν 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμό 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος προϋπολογισμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προϋπολογισμών 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά Πρέπει να σηκώνετε το χέρι σας παρακαλώ. Ξανά, τρία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, τέσσερα, πί. α, τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα, τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε σας παρακαλώ, συνάδελφοι. Δεν ψηφίζετε. Πέρας ψηφοφορίες. 42 υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 5 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν. And, uh, the last vote... Τελευταία ψηφοφορία τώρα το πρωί, ενδεικτική ψηφοφορία για την ε, πρόταση κανονισμού Συμβουλίου και, ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την περίοδο 2014-2020 του κατάρτιση του προγράμματος Δικαιώματα και Ιθαγένεια. Η κυρία Γκέντς θέλει να λάβει το λόγο, η συγγήτρια. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα ευχαριστώ όλους που συνέβαλαν. Τις ε, πέντε επιτροπές που γνωμοδότησαν ε, η Επιτροπή Απασχόλησης που συνεργάστηκε με τον κανονισμό 50. Ήταν περίπλοκο και καθόλου εύκολο να βρεθούν ισορροπίες, αλλά νομίζω ότι θα είναι ισχυρό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με Συμβούλιο και Κομισιόν. Ευχαριστώ και πάλι όλους που συνέβαλαν. Ευχαριστώ κυρία Γκέντσι. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Ε, προϋπολογισμού 1. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Προϋπολογισμού 2 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 21, την Επιτροπή Γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 112 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε έλεγχος ηλεκτρονικός ψηφίζουμε την 112 άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 26 υπέρ 24 κατά χωρίς αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 6 σε δύο τμήματα, τμηματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προπάμε στη συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. στην 26. Ψηφίζουμε μόνο ένα μέρος της υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι, α, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ΦΑΜ 26, ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. 19 υπέρ, 29 κατά, 2 αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έλεγχος ηλεκτρονικός ΦΑΜ 29 από την Επιτροπή Γυναικών. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 27 υπέρ 22 κατά, μία αποχή δεκτή. Πάμε τώρα στην συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Employment 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 140 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ, σηκώνετε το χέρι σας. Κατά 140. Ψηφίζουμε ξανά υπέρ. Κατά. Αποχές. Λοιπόν, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 140. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 18 υπέρ 19 κατά 13 αποχές. Ε, 5 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμ... 525 25, Επιτροπή Αναφορών υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Employment 22, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 527, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 18, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 19 υπέρ, κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 19. ΦΑΜ 38, ένα μέρος μόνο υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 40 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβιβαστική 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά φαμ 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 164 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, budget 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 173 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Employment 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Budget 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 184 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 41 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 42 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 43 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, ΦΑΜ 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πάμε τώρα σε αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές. 49 ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 52 και budget 3. Α, δεν είναι παραδεκτές. Πάμε στη 46. Υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 31 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Employment 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Employment 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΑΜ 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΦΑΜ 9 ε, ναι, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ 83 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ψηφίζουμε την τροπολογία 83 γιατί δεν βλέπω τα χέρια να σηκώνονται Α, μισό λεπτό να τελειώσουμε την ψηφοφορία στην 83. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 83 δεν ήταν σαφές. Ψηφίστε παρακαλώ. Συνάδελφοι, πέρα της ψηφοφορίας. 20 υπέρ 30 κατά, άρα απορρίπτεται και πάω πίσω στη ΦΑΜ 11 γιατί το προσπέρασα κατά λάθο. ΦΑΜ 11 υπέρ κατά εποχές ε, απορρίπτεται και συνεχίζουμε με τη συμβιβαστική 34 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 36 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, budget 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά πρέπει να κάνουμε έλεγχο στην 13 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. 28 υπέρ, 23 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία 38. Ποιο είναι υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 98. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 40, συμβαστική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 και τη Επιτροπή Απασχόληση 12. Ποιο είναι υπέρ, είναι πανοπιότυπε. Κατά αποχέ εγκρίνονται. 15 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 41 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 17 τη Επιτροπή Γυναικών υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της Επιτροπής Γυναικών κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει, ψηφίζουμε το δεύτερο μόνο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19 των γυναικών υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβεστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 της Επιτροπής Απασχόληση, υπέρ κατά δεν βλέπω διαφορά, δεν σηκώνατε τα χέρια. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Ψήφισαν 30 υπέρ, 20 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. 20 γυναικών υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. ψηφίσατε. Τέλος. Ψήφισα 47 υπέρ, 2 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Γκέντς. Και ολοκληρώσαμε. Εγκαίρος. Ή όχι. Α, όχι, λάθος. Έχουμε και άλλη ψηφοφορία, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν τελειώσαμε. Θα πρέπει να υποβάλουμε σύσταση προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για, την, ε, για τον ορισμό δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με ειδικέ γνώσεις στον τομέα ναρκωτικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας που εδρεύει στη Λισαβόνα με βάση τους κανόνες της διάσκεψης των Προέδρων. Παρακαλώ, συνάδελφοι, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών πρέπει να εγκρίνει ένα κατάλογο με υποψηφίους που είναι επιλέξιμοι για το διορισμό. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά, διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλον και οι ψήφοι υπέρ θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη ε, της επιστολής με τους προτινόμενους υποψηφίους προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεν θα γίνουν δεκτές ούτε αρνητικέ ψήφοι ούτε εποχέ. Μόνο οι ψήφοι περ υπολογίζονται. Μετά την έκβαση ψηφοφορία, ο κατάλογο των υποψηφίων θα καταρτιστεί με βάση τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. Για τις πρώτες δύο θέσεις ε, θα προτείνουμε τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και για την τρίτη και τέταρτη θέση θα προτείνουμε ε, για τους αναπληρωτές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης. Οι πολιτικές ομάδες πρότειναν πέντε υποψηφίους. Θα τους αναφέρω με αλφαβητική σειρά. Ακούστε παρακαλώ. Mr. Massimo Cano, proposed by EP. Massimo Cano από το ΕΛΚ. Καρμέλα Κώστα από το ΕΛΚ πρόταση. Μπαρ Παρατούρκο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Καταλά Φελίντσι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κάρλα Ρώση από την Άλντε. Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά τις υποψηφιότητες με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως σας είπα και προηγουμένως. και θα πρέπει να κληρώσουμε με ποιο όνομα θα ξεκινήσουμε και κατόπιν θα ακολουθήσουμε την αλφαβητική σειρά. Επιλέγεται ο κύριο Μασίμο Κάνο. Α, εντάξει, ούτως ή άλλως στηρείται η αλφαβητική Ξεκινάμε. Ψηφίζουμε ξεχωριστά, επαναλαμβάνω, τους υποψηφίους. Και το Μάσιμο Κάνο πρώτη ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είναι πρόταση του ΕΛΚΟ, κύριος Μάσιμο Κάνο. Παρακαλώ ψηφίστε ηλεκτρονικά. Δεύτερος στο κατάλογο. Είκοσι ψήφους ε, υπέρ έλαβε ο κύριος Κάνο. Η κυρία Καρμέλα Κώστα τώρα. Ψηφίζουμε για την κυρία Καρμέλα Κώστα πρόταση του ΕΛΚ, υποψηφιότητα της κυρίας Κώστα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. κυρία Κώστα συγκέντρωσε 19 ψήφους. Μπάρμπαρα Ντούρικοπ Ντούρικοπ, πρόταση των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Yes. 34. 34 ψήφου συγκέντρωση, η κυρία Ντύρκοπ. Force, Mrs. Katalin. Καταλήν Φελβίντσι. Πρόταση των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Ψηφίζουμε. Close the vote. Τέλος ψηφοφορίας, 21 ψήφους έλαβε η κυρία Βίτση και η κυρία Κάρλα Ρώση, πρόταση των ε, φιλελευθέρων. Ψηφίζουμε, παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 31 ψήφους Η κυρία Ντύρκο Πτύρκο συγκέντρωσε 34 ψήφου, είναι πρώτη στο κατάλογο. Η κυρία Καρλαρώση δεύτερη με 31 ψήφου. Αυτέ είναι οι δύο προτάσει για, για τους ανεξάρτητου Τρίτη είναι η κυρία Καταλήν Φαλβίντσι, 21 ψήφου. Και ο κύριο Μάσιμο Κάνο, 20 ψήφου, είναι ο τέταρτος. Οι δύο τελευταία θα είναι οι προτάσει για αναπληρωτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε με τη συνεδρία των συντονιστών σε μισή ώρα, λέει η Πρόεδρος.